Okay, colleagues, people can start taking their... Συνάδελφοι, μπορείτε να αρχίσετε να τακτοποιήσετε. Είναι μεγάλη συνεδρίαση, θα κρατήσει πολύ, το ίδιο και η ψηφοφορία. Και για πρώτη φορά έχουμε τρεις επιτροπές που συνεργάζονται για ένα θέμα συναπόφασης. Η κάρτα μου δουλεύει επιτέλου, Η δική μας Επιτροπή ε, ε και άλλες δύο επιτροπές, ΑΦΕΤ και ΜΠΟΥΤ, να ξεκινήσει λοιπόν η κοινή αυτή συνεδρία των τριών επιτροπών. Έχουμε τρία σημεία στην ημερήσια, τέσσερα μάλλον σημεία στην ημερήσια διδαξή μας. Το πρώτο έγκριση αυτής. Δεν ζητήθηκαν αλλαγέ. Μπορούμε να την εγκρίνουμε όσο έχει. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν έχω ανακοινώσει υπό το σημείο 2. Αλλά για τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, κοινή συνεδρία 28 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου, βρίσκονται στου φακέλου σα. Σημείο 3. Εάν έχετε παρατηρήσει, παρακαλώ να ειδοποιήσετε τη γραμματεία στο τέλο τη συνεδρίαση. Ιδάλω θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 4. Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΤΒΑ, για τη δημιουργία των εγγύσεων ΕΤΒΑ και Ταμείο Εγγύσεων ΕΤΒΑ. Τρεις συνεισηγητές. Μου είπαν και οι τρεις ότι δεν ε, επιθυμούν να λάβουν το λόγο σε αυτή τη φάση. Οπότε μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ε, ψηφοφορία. Πριν από αυτό όμως θέλω να καλωσορίσω έναν ειδικό προσκεκλημένο σήμερα το Λόρδο Μάρλαντ. Κάθεστε πίσω, Λόρδε, πρόεδρος του ε, Συμβουλίου ε, Επενδύσεων και Επιχειρήσεων της Κοινοπολιτείας από το Εμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Λοιπόν, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Πριν ξεκινήσει, να κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Πατήστε ό,τι κουμπί σας αρέσει μόλις ε, αρχίσει η ψηφοφορία. Άρχεται. Has everybody voted? Εψήφισαν άπαντες. Δεν ψήφισαν όλοι. Εάν θέλετε να ψηφίσετε, δείτε αν λειτουργούν οι κάρτες σας παρακαλώ. Τέσσερις δεν ψήφισαν. Εάν θέλετε να σας βέβαιοι ότι λειτουργούν τα μηχανήματα οι κάρτες, ψηφίστε. Σχεδόν τα καταφέραμε. Κάποια τώρα έβαλαν τις κάρτες στα μηχανήματα. Κυρία Τόγια, δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Καπιανού δεν λειτουργεί το μηχάνημα ή δεν έχει βάλει την κάρτα του ένας, ένας συνάδελφος. Εκτός και αν θέλετε να μην ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ωραία. Όλα πάνε καλά, λειτουργούν τα μηχανήματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Έχουμε μια μακρά ψηφοφορία με 22 συμβαστικέ. 22 είναι. Όχι, 25. 25 είναι συμβαστικέ, τι έχετε δει και ελπίζουμε ότι θα διευκολύνουν την ε, ψηφοφορία μα. Ευχαριστούμε του συνεισηγητέ για αυτήν την ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την 71. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίβεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Αγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. Προφορική τροπολογία από το συντάκτη για το άρθρο 197. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Άρχεται η προφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 222. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 222. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη. Και είναι και ευκαιρία να ξυπνήσουν όλοι. Πέρας. Ναι, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Παρακαλώ να σηκώνετε λίγο τα χέρια σας. Διότι είναι τεράστια η αίθουσα, δεν βλέπω τόσο καλά μακριά. 30. Α, καταπίπτει. 223, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Έλεγχος. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος, ε, ε, τροπολογία ελέγχων του προπολογισμού 14. Υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 14, άρχεται την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται δίκιο είχατε που θέλατε να ελεγχθεί.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 είναι ταυτόσιμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 271. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν παντέ πέρα Εγκρίνονται. Καταπληκτούν. 274 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. 39 υπέρ. Α, και αυτή καταπίπτει. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για να πάμε σε μια σελίδα παρακάτω. 10 στο δικό μου κατάλογο, σελίδα 10. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έλεγχος προφορικής τροπολογίας 1. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Κόντ 16 και κόντ 27 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 381. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος στις 381. Άρχεται η ψηφοφορία. αν ανάπαντες. Πέρας. Απορρίπτονται. 293 υπέρ. Έχω κάτι πολύ περίπλοκες εξηγήσει εδώ για το τι γίνεται με τον κατάλογο. ...293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά από μακροσκελή συζητήσεις. 294 με προφορική τροπολογία τη συντάκτη. Τη συντάκτρια. Υπέρ, κατά, εποχέ. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε το 294 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Άρχεται του ψηφοφορία μάλλον. Ψήφισαν άπαντε. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Και πάλι, η 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 295 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έλεγχος στις 295, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 305 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 307. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για 309 Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχο 412. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 313 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για την 313 να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 314 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 317 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 318 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τα 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τα 221 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έλεγχος για το 221 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνονται. 53 υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε, Τα 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο για την 320 έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Όχι. Λίγο χρόνο. Εψήφισαν άπαντες τώρα. Πέρας της ψηφοφορία, Απορρίπτεται 54, σωστά. 54 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 323 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισε να απαντές πέρα της ψηφοφορίας. Απολύπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνονται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη 325. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνονται. 324. Με συγχωρείτε, 327. 327 ε, υπέρ, κατά, αποχέ να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 327. Εψήφισαν ε, άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 329 και 330 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 334 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 335 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 336 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 337 και 339 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. 338 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 340 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 341 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κόντ 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κοντ 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 364. Καταπίπτει. 365 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχο. Έλεγχο για την 365. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτω. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 372. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύπτω. 375 υπέρ κατά εποχές. Ελέγχουμε για το 375 άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 276 και 42 από την κοντ μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 ελέγχου είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 44 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται με μια ψηφοδιαφορά. Πολύ μικρή διαφορά. 45 από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού υπέρ κατά αποχέ, Να ελέγξουμε για την κόντ 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 378 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 έλεγχο των προπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 380. 380 ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Κοντ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 382 υπέρ. Κατά. απόχέ Να ελέγξουμε για τα 382. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας, απορρίπτεται. 385 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά δεν εγκρίνεται. 93 και 94 και 95 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 97 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, έλεγχος για την 97. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενενήντα οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Του κυρίου Ντέβα, του αντιπρόεδρου μας. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύτωτα. 100 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Ή 103 λέει. Θα πηδήξουμε ώστε την 103. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος. Έλεγχος για την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Επίσης ανάπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. 109, ναι. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. Με τεράστια διαφορά. Με συγχωρείτε. Μερικοί κουράστηκαν. 21. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε βγάλει τα τρίτα τέταρτα του καταλόγου. Συνοδεύει. Φουράγιο. 111 και 172 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Να ελέγξουμε. έρχεται η ψηφοφορία. 111 και 172 από κοινού. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Οι 6 και 20. Οι άλλε καταπληκτούν. Όχι, και αυτέ καταπληκτούν. 173. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. 173 άρχεται ψηφοφορία. Εξής, ανάπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 174 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό. Όχι. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 8. Καταπίπτει. 118 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 9. 10 Συγγνώμη. 10 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Κον 420 ταυτόσιμε από κοινού υπέρ κατά αποχέ. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε για αυτέ Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτωτο. Απορρίπτωτο. Να κάνουμε έλεγχο μου λένε. 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, μερικοί καθυστέρησαν να κουνήσουν τα χέρια τους. Ε, εψήφισαν άπαντες όσοι έπρεπε να ψηφίσουν. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 129. ξανά πάντα πέρα τη προφορία. Αγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν βλέπω να κάνετε κάτι εκεί. Ξανά. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Αγκρίνεται. 135 Τεκώνεται 7 από κοινού υπέρ κατά εποχές έλεγχος. Έλεγχος 135 και κόλτα αυτά άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Και εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω τους σοσιαλιστές. 136 ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισε να απαντήσω. Πέρας. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. αποχέ. Έλεγχος για τον 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141-142 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος για τα 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ξεχωριστέ ψηφοφορίες 148 Κατά τμήματα μάλλον. Πρώτο τμήμα. Με προφορική τροπολογία για την 148. Υπέρ. Κατά αποχέ. Απολύτω. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχέ. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 149 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Κόρτ 8. Καλύπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 151, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, έχει και προφορική τροπολογία μαζί. 163 με την προφορική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164. Καταπίπτει. Και άλλη καταπίπτει. 165 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Για να ξαναπάμε. 165 υπέρ. Κατά. εποχέ, Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 165. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Εποχέ να ελέγξουμε για την 166, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Κοντ 10. πέρα, Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε την 167. Άρχεται η ψηφοφορία. Εύσεις ανάπαντες πέρας. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ελέγξουμε για την 168. Άρχεται ψηφοφορία. Έψηφες ανάπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Σχεδόν τελειώσαμε. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Εποχές. Για να ελέγξουμε για την 178. άρχιτε ψηφοφορία. Εψήφισαν ανάπαντες για την 178. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν ανάπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στους τρεις συνεισηγητές. Μπράβο σας. Μην φύγετε όμω. Συνάδελφοι, μην φεύγετε. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Κύριε Φρουτζουλίτσα, θέλετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, ε, τους βουλευτές που παρευρίσκονται σήμερα εδώ ε, και ψήφισαν αυτήν την, υπερψήφισαν μάλλον την πολύ σημαντική έκθεση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Και αυτό γιατί είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τρει συνεισηγητέ, αλλά και επειδή εδώ αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο θα αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ε, βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και των Αφρικανικών χωρών αλλά και των χωρών της ε, Ανατολικοευρωπαϊκής Γειτονίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το προωθεί γενικά την ανάπτυξη και τη σταθερότητα σε όλες αυτές τις περιοχές ε, του κόσμου και αποτελεί βέβαια ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο της ήπιας ισχύω soft power της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίησή του καταδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει ε, στη θέση που έχει σήμερα ως ένας σημαντικός παγκόσμιος ε, παίκτης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, θα ψηφίσουμε τώρα επί της απόφασης του να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή έναρξη του τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε 72 ψήφους ε, για να εγκριθεί αυτή η απόφαση. Οπότε ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Some people haven't voted yet. Κάποιοι δεν έχετε ψηφίσει ακόμα. Πρόκειται για σημαντική ψηφοφορία. Αν θέλετε να ξεκινήσει ο τριμερούς διάλογο πρέπει να ψηφίσετε. Έχετε λοιπόν ψηφίσει όλοι. Άπαντες. Υπάρχει κάποιος χωρί κάρτα. Καλώ έβαλε και ο συνάδελφο εδώ. Την κάρτα στο μηχάνημα. Καλώς. Πέρασε λοιπόν τη ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν καταφέραμε την πλειοψηφία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε λοιπόν τους εισηγητές. Ε, και προφανώς επειδή ε, έχουμε τρεις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές που συμμετέχουν εδώ θα πρέπει βέβαια να μοιραστούμε μεταξύ μας τις αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή μας στον τριμερή διάλογο. Θα το κανονίσουμε βέβαια αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και καλό απόγευμα.